Σας καλωσορίζω στην ε, πρώτη κοινή συνέλευση Envy και Ντέβε σχετικά με τους ε, στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Ε, θα ήθελα να καλωσορίσω τον Επιτροπό Μίμητσα που θα μας ενημερώσει πάνω στην πρόοδο που έχει σημειωθεί. Όσον αφορά τα πρακτικά θέματα, θα κάνουμε το εξής. Επειδή ο Επίτροπος έχει μέχρι τις 6 η ώρα ε, ώρα στη διάθεσή του, θα πρέπει να εργαστούμε αποτελεσματικά. Θα ακολουθήσουμε τη διαδικασία catch the eye. Όποιος θέλει να θέσει ερώτηση θα πρέπει ε, να σηκώσει την ταμπελίτσα του, ώστε να γνωρίζουμε ποιος θέλει να θέσει ερώτηση. Θα καταρτήσουμε κατάλογο των ομιλητών και ελπίζουμε όλοι να μπορέσετε να πάρετε το λόγο, αλλά αυτό βέβαια θα εξαρτηθεί από το χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας. Ε, υπολογίζουμε ότι θα προλάβουμε να ακούσουμε 15 με 20 ερωτήσεις. Ένα λεπτό θα έχει ο καθένας στη διάθεσή του. Σας παρακαλώ λοιπόν, προετοιμάστε την ερώτησή σας καταλήλως. Πρόκειται για την πρώτη κοινή μας ε, συνεδρίαση όπου παρακολουθούμε την, ε, εκτέλεση, την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης και του θεματολογίου 2030. Ε, ο ε, ε, Αντιπρόεδρος Τίμερμαν της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παρουσίασε το έγγραφο προβληματισμού και ακούσαμε και στοιχεία σχετικά με την έκθεση για τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης και μετά από την ακρόαση αυτή το Κοινοβούλιο υιοθέτησε τον Μάρτιο του 2019 ψήφισμα για, τα, για τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, ε, όπου ε, εκφράζεται υπέρ του εγγράφου προβληματισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, ζητάει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει μια γενική, μια συνολική στρατηγική για την επίτευξη των στόχων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη, που να συμπεριλαμβάνει και εσωτερικές και εξωτερικές πολιτικές. Κύριε Επίτροπε, περιμένουμε να ακούσουμε την παρουσίασή σας πρώτα όμως θα ήθελα να δώσω το λόγο στον ε, αγαπητό μου συνάδελφο, τον ε, Τόμας Τομπέ, που είναι πρόεδρος της Επιτροπής Ανάπτυξης. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Έικχαουτ. Θα ήθελα και εγώ να πω ότι είναι πολύ ωραίο που ξεκινάμε την κοινοβουλευτική μας ε, θητεία με κοινή συνεδρίαση των επιτροπών μας και μάλιστα παρουσία του Επιτρόπου. Θα ήθελα να δράξω την ευκαιρία να πω ότι είναι σημαντικό για τις δύο επιτροπές μας να επιδείξουμε ηγετικό ρόλο εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ώστε να διασφαλίσουμε την πλήρη εφαρμογή των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης στις ευρωπαϊκές πολιτικές. Όπως γνωρίζετε, ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών τόνισε ότι παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί σε μια σειρά τομέων τα τελευταία τέσσερα χρόνια όσον αφορά τους στόχους. Ε, όσον αφορά κάποιους στόχους ήταν πολύ αργή η, η πρόοδος ε, ή έχει ε, αντιστραφεί η πρόοδος. Ε, μετά από την ε, πρώτη Σύνοδο Κορυφή για του Στόχου Βιώσιμη Ανάπτυξη το 2015, οι δύο επιτροπέ μα που ήταν παρούσες και στην διάσκεψη έχουν παρακολουθήσει το θέμα και γι' αυτό χαίρομαι που ο επίτροπο Μίμητσα θα μας παρουσιάσει σήμερα μια επισκόπηση που συμπεριλαμβάνει και την ε, κοινή έκθεση για την ε, επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξη σε όλον τον κόσμο. Είναι κοινή έκθεση διότι τονίζει τι δράσει και των κρατών μελών ε, και τη Ευρωπαϊκή Ένωση. όσον αφορά μάλιστα τη βοήθειά μα προ αναπτυσσόμενες χώρε για την επίτευξη των στόχων. Θα παρακαλούσα λοιπόν τον Επίτροπο Μίμητσα να μα ενημερώσει και σχετικά με τη διάσκεψη κορυφή του Σεπτεμβρίου. Παρακαλώ. Σας ε, ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα αξιότιμοι ευρωβουλευτές. Ε, σας καλωσορίζω θερμά τώρα στην έναρξη της νέας κοινοβουλευτικής θητείας. Καλωσορίζω λοιπόν ε, όλα τα μέλη της Επιτροπής ΕΝΤΕΒΕ και της Επιτροπές ΕΝΒΗ και καλή επιστροφή θα ήθελα να πω στους, στους επιστρέφοντες. Η εφαρμογή του θεματολογίου για τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης είναι ένα από τα πιο σημαντικά με τα οποία θα, ασχοληθεί, ε, θα ασχοληθούν οι επιτροπές σας τα επόμενα χρόνια. Ελπίζω να μπορώ να σας δώσω μια καλή επισκόπηση ε, του ε, Υψηλού Πολιτικού Φόρουμ της προηγούμενης εβδομάδας και να σας βοηθήσω να προετοιμαστείτε για τη διάσκεψη κορυφή το Σεπτέμβριο στη Νέα Υόρκη όπου θα συμμετάσχουν αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων. Το θεματολόγιο 2030 αποτελεί σημαντική μετάβαση όσον αφορά τον τρόπο που προσεγγίζουμε την ανάπτυξη. Διότι ξεπερνάει το θέμα της κρίζωσης της στόχιας, καλύπτει όλες τις πτυχές βιώσιμης ανάπτυξης, ε, κοινωνικές, ε, οικονομικές και περιβαλλοντικές πτυχές και ισχύει για όλες τις χώρες ε, και εντός του Ευρωπαϊκού, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έπαιξε σημαντικό ρόλο στην κατάρτιση του θεματολογίου και παραμένουμε αποφασισμένοι να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να προωθήσουμε την εφαρμογή του θεματολογίου και στις πατρίδες μας και στον υπόλοιπο κόσμο. Φέτος κλείνει ο πρώτος τετραετής κύκλος του Φόρουμ και τον Σεπτέμβριο θα ξεκινήσει η ε, αναθεώρηση, η επισκόπηση και η προηγούμενη εβδομάδα ε, έθεσε το πλαίσιο για τη συνάντηση του ε, ε, Σεπτεμβρίου. Ένα θετικό σημάδι ήταν ότι το σχέδιο της πολιτικής διακήρυξης, ε, το αποτέλεσμα δηλαδή της διάσκεψης του Σεπτεμβρίου συμφωνήθηκε από όλα τα κράτη του ΟΗΕ ήδη πριν ε, την πραγματοποίηση του φόρουμ του Ιουλίου. Αυτό δεν ήταν ε, αυτονόητο δεδομένων των προκλήσεων που έχουμε αντοπίσει στο παρελθόν για την επίτευξη για την συμφωνία πάνω σε κείμενα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έπαιξε σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του κειμένου. Είναι ένα εστιασμένο κείμενο που περιλαμβάνει χρήσιμες διατυπώσεις για κάποιες από τις βασικές μας προτεραιότητες, ισότητα, κλίμα, ε, περιβάλλον, ε, πολυμέρεια, παρακολούθηση δεδομένων και αξιολόγηση. Θα θέλαμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη διακήρυξη για να προωθήσουμε πιο γρήγορες δράσεις ε, όσον αφορά του στόχου βιώσιμης ανάπτυξης του τους επόμενους μήνες και τα επόμενα χρόνια. Και ελπίζω εσείς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μπορέσετε να μας βοηθήσετε στην προσπάθεια αυτή. Ε, τα Ηνωμένα Έθνη θα ήθελαν να ξεκινήσουν μια δεκαετία δράσεων ε, για το, την επίτευξη των στόχων βιώσιμη ανάπτυξη το Σεπτέμβριο. Στην δήλωση που έκανα στο όνομα τη Ευρωπαϊκή. Ευρωπαϊκής Ένωση και των ε, κρατών μελών. Τόνισα τη δέσμευσή μα ε, να πετύχουμε ε, τους στόχους του θεματολογίου 2030. Οι 26 από τα 28 μας κράτη-μέλη ήδη έχουν υποβάλει τις εθελούσιες εθνικές ανασκοπήσεις το γεγονό αυτό είναι πολύ θετικό και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη παρουσιάσει τα δικά τη αποτελέσματα τη παρακολούθηση. Ο Επίτροπο Βέλα και εγώ ε, οργανώσαμε μία επιμέρου εκδήλωση μαζί με τη Φιλανδική Προεδρία του Συμβουλίου για να τονίσουμε τι δράσει που έχει αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη για την εφαρμογή των στόχων βιώσιμη ανάπτυξη και εσωτερικά και εξωτερικά. Ε, ένα πράγμα ήταν σαφές ε, από την αρχή. Ο κόσμος περιμένει από εμά να αναλάβουμε ηγετική θέση στις ε, παγκόσμιες προσπάθειες για εφαρμογή του θεματολογίου του 2030. Η εκδήλωση αυτή προσέλκυσε το ενδιαφέρον πολλών και επενέθηκε από πολλούς συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Εθνών και του Γενικού Γραμματέα τους. Μπορέσαμε να επιχειρηματολογήσουμε υπέρ της Ευρώπης ως πρωτοπόρου ε, στην βιώσιμη ανάπτυξη. Είχαμε λοιπόν το έγγραφο προβληματισμού προς ε, μια ε, βιώσιμη Ευρώπη 2030 που εκδώσαμε ε, φέτος. Εδώ καθορίζονται προτεραιότητες για το πώς θα προχωρήσουμε και πώς θα πετύχουμε την μετάβαση σε μια βιώσιμη Ευρώπη και πώς θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια πλήρως κυκλική οικονομία, πώς θα μπορέσουμε να έχουμε πράσινη ενέργεια και μεταφορές και πώς θα μπορέσουμε να ενισχύσουμε τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και να χρησιμοποιήσουμε εργαλεία πολιτικής όπως είναι η εκπαίδευση, ε, η ψηφιοποίηση, η χρηματοδότηση και η φορολογία για να πετύχουμε του στόχου αυτού. Επίση έχουμε την έκθεση προόδου για του στόχου βιώσιμη ανάπτυξη που εκδόθηκε από τη Eurostat τον Ιούνιο που επιβεβαιώνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σημειώσει πρόοδο ε, σχεδόν ε, σε όλου του στόχου. Αν και σε μερικού η πρόοδο ήταν πιο αργή από ότι ε, σε άλλου. Ιδιαίτερα όσον αφορά κάποιου περιβαλλοντικού στόχου, απαιτούνται περισσότερες προσπάθειες. Επίσης έχουμε την έκθεση 2019 για την πολιτική σύγκληση που δείχνει πώς οι ευρωπαϊκές πολιτικές λαμβάνουν υπόψη τον πιθανό αντίκτυπο σε αναπτυσσόμενες χώρες. Και τέλος είχαμε την πρώτη ε, συνολική έκθεση για την εφαρμογή της ε, ε, συνένεσης του 2017 για τις προσπάθειες ε, για τους ε, στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Ε, εξετάζουμε την κατάσταση και στις χώρες εταίρους μας. Η συνένεση αυτή έχει αναγνωριστεί ως σημαντική συμβολή στην, επίτευξη του, στην εφαρμογή του θεματολογίου 2030 σε παγκόσμιο επίπεδο. Και είμαι ευγνώμων προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που συνεργάστηκε μαζί μας και με το Συμβούλιο για να τα τα καταστήσει όλα αυτά δυνατά έτσι έχουμε ξεκινήσει κάποιες νέες δράσεις όπως είναι η Συμμαχία Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αφρικής ε, ή ε, το σχέδιο ε, εξωτερικών επενδύσεων όπου προβλέπεται η κινητοποίηση 44 εκατομμυρίων ευρώ για επενδύσεις στην Αφρική. Επίσης, στο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο προβλέπονται σημαντικές επενδύσεις. Σε συνεργασία με πολυμερείς οργανισμούς και ιδιαίτερα με τα Ηνωμένα Έθνη, όπως άλλωστε φαίνεται και από την πρωτοβουλία Spotlight ε, ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ για να δοθεί τέλος ε, στη βία εις βάρος ε, γυναικών και κοριτσιών. Ε, Ήταν πολύ ενδιαφερόμενοι φορείς ε, παρόντες ε, στην εκδήλωση που οργανώσαμε. Εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών, του ιδιωτικού τομέα και του πανεπιστημιακού χώρου. Θα πρέπει όμως να δείξουμε ότι εφαρμόζουμε ενεργά τους στόχους για να εμπνεύσουμε και άλλους να εφαρμόσουν τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Και για να είναι βιώσιμη η ανάπτυξη, θα πρέπει να σκεφτούμε ότι όλοι είμαστε αναπτυσσόμενες χώρες, όλοι έχουμε πράγματα που πρέπει να κάνουμε. Θα πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειες για θετικές δράσεις ε, για να έχουμε βιωσιμότητα σε όλα τα, σε όλους τους τομείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ούρσουλα Φοντερ Λάγεν, ε, που εξελέγει πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την προηγούμενη εβδομάδα τόνισε την ανάγκη ε, τόνισε πόσο σημαντική είναι η στόχη βιώσιμης ανάπτυξης ε, και πόσο σημαντικό είναι το ευρωπαϊκό εξάμεινο για να ε, μπορέσουμε να διατηρήσουμε τις προσπάθειές μας. Είναι πολύ σημαντική η πρόταση αυτή και ελπίζω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να τη στερέξει. Σε εξωτερικό επίπεδο θα πρέπει να βρούμε νέα χρηματοδοτικά μέσα για την βιώσιμη ανάπτυξη και θα πρέπει να τα λάβουμε όλα αυτά υπόψη στη μελλοντικό μας προγραμματισμό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο σημαντικότερος παράγοντας ε, ε, ε αναπτυξιακής βοήθειας σε όλο τον κόσμο και παρέχει 75 δισεκατομμύρια ε, ευρώ για τέτοιες δράσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη της Είμαστε ο μεγαλύτερος παράγοντας παγκοσμίω στο χώρο αυτό. Η επίσημη ανακτησιακή βοήθεια ε, αποτελεί το βασικό μας χρηματοδοτικό όργανο, ε, κυρίως για την κρίζωση της στόχιας σε παγκόσμιο επίπεδο και ιδιαίτερα στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες ε, και σε έθραυστα περιβάλλοντα. Αλλά η προσπάθειε μας όσον αφορά τους στόχου βιώσιμη ανάπτυξης ε, δεν επικεντρώνονται αποκλειστικά στην ε, επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια. Κινητοποιούμε ε, δημόσιους και ιδιωτικούς πόρους και πιο σημαντικό είναι ότι δεν προσπαθούμε απλά να είμαστε ο πιο σημαντικός παράγοντας στον τομέα αυτόν σε όλο τον κόσμο. Θέλουμε να είμαστε ο καλύτερο. Και αυτό σημαίνει να ε, δημιουργήσουμε εταιρικέ σχέσεις με όλους τους άλλους εταίρους μας στο θεματολόγιο ε, για τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης και το 2030. Θα πρέπει να παραμείνουμε ισχυροί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα πρέπει ε, η κλιματική μας και αναπτυξιακή μας δράση να ευθυγραμμίζεται με μια προσέγγιση που να βασίζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα, που να έχει στόχο την πολιτική συνοχή στην ανάπτυξη, την σύγκληση ε, και την πολιτική ειρήνης και ασφαλείας. Στο περιθώριο του Φόρουμ ε, Υψηλού Επιπέδου συζητήσαμε με τους εταίρους μας ε, πώς μπορούμε να επιταχύνουμε την εφαρμογή των στόχων ε, βιώσιμη ανάπτυξης. Εξετάσαμε θέματα χρηματοδότησης και παρακολούθησης. Παρουσιάσαμε την έννοια ολοκληρωμένων πλαισίων χρηματοδότησης ε, ώστε να κινητοποιήσουμε ε, πόρους όλων των ειδών εθνικών, διεθνών, δημοσίων και ιδιωτικών. Το φόρουμ αυτό επίσης μου έδωσε μια ευκαιρία να έχω μια σειρά διμερών συναντήσεων για παράδειγμα, ε, και με τον ε, παλαιό και με τον νέο ε, πρόεδρο του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας του ΦΑΟ. Επίσης, με τη Γαλλία, την Ισπανία και το Μεξικό εξετάσαμε τη σχέση ανισοτήτων και αλλαγής του κλίματος. Στόχος μας είναι να αντιμετωπίσουμε την ανισότητα σε όλες ε, τις διαστάσεις της. Ε, ελπίζω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συνεχίσει να επικεντρώνεται, να εστιάζει στο θέμα αυτό κατά τη διάρκεια του της συστητίας. Κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτές, ε, έχουμε ένα τεράστιο έργο μπροστά μας. Το νέο Κοινοβούλιο και η Νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, θα έχουν σημαντικές ευκαιρίες να επιταχύνουν τις εργασίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, όσον αφορά του στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Ε, θα ήθελα να επικρατήσω τις προσπάθειες και των δύο επιτροπών σας κατά την προηγούμενη θητεία για απλοποίηση και εφαρμογή του θεματολογίου για τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Προσβλέπουμε στη στενή συνεργασία μαζί σας τους επόμενους μήνες και τα επόμενα χρόνια και προσωπικά προσβλέπω στο να ξανασυναντήσω όλους σας το Σεπτέμβριο στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Thank you very much. So we now do... ο πρώτος γύρος ερωτήσεων. Ένα λεπτό θα έχει ο καθένας, ε, ώστε να έχουμε στο δυνατόν περισσότερους να πάρουν το λόγο. Συνάδελφος Μπουζόη είναι ο πρώτος από το ΕΛΚ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε αγαπητέ Επίτροπε. Δεν είναι αυτό ο σκοπό οι στόχοι βιώσιμη ανάπτυξη, όπω υπόθηκε, όμω θα μα βοηθήσουν να βελτιώσουμε τον κόσμο. Είναι 17 οι στόχοι, θα εστιάσω στον υπαριθμό 3, που έχει άμεση σχέση με την υγεία. Φυσικά και εδώ τα πάμε καλύτερα από άλλε του κόσμου. Σε παγκόσμιο επίπεδο γίνανε πρόοδοι τα τελευταία χρόνια, λιγότεροι παιδικοί θάνατοι, ε, εν πολλής λόγω των εμβολιασμών. Επίσης έχει πέσει και η θνητότητα των ε, νεαρών μητέρων, έχει πέσει ο ε, του ιούδου του AIDS λόγω των αντιρρετροϊκών φαρμάκων Επίσης, αλλονοσία και φυματίωση είναι σε ύφεση, όμως η φυματίωση εξακολουθεί να είναι ένα πρόβλημα, όχι μόνο σε άλλες υπήρους, αλλά και σε κάποιες ε, χώρες της κεντρικής και ανατολικής και νότιας Ευρώπης. Το ερώτημά μου, αφού πω βέβαια ότι πρέπει να βελτιώσουμε και τους στόχους μας και την κατάσταση, το ερώτημά μου είναι πώς μπορούμε να συνεισφέρουμε στην επίτευξη του στόχου παριθμών 3 σε παγκόσμιο επίπεδο. Ευχαριστώ. Thank you very much. Σας ευχαριστώ. Δεύτερη ερώτηση από τους σοσιαλιστές και δημοκράτες, ο κύριος Μπούλμαν. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε μη αν με επιτρέπετε, θέλω να σας ευχαριστήσω για ό,τι κάνατε, γιατί το προηγούμενο κοινοβούλιο ε, σας είναι ευγνώμων για τον τρόπο με τον οποίο πιέσατε για τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης και σήμερα μας δώσετε ένα μάθημα ακόμα για το τι πρέπει να γίνει τους επόμενες μήνες και τα επόμενα χρόνια. Μια ερώτηση. Βρισκόμαστε εν, μέσω, εν μέσω μιας ολιστικής άσκησης εμπόριο και αναπτυξιακή πολιτική συνδυάζουν διάφορα στοιχεία της πολιτικής σφαίρας, γεωργία, περιβάλλον, κοινωνική πολιτική, οικονομική πολιτική. Και πώς μπορούμε να συσχετίσουμε όλες τις προσπάθειες βελτίωσης κατάστασης με το κρίσιμο ζήτημα των ανισοτήτων που αναφέρατε και πολύ σωστά οι ανισότητες είναι το βασικό εμπόδιο κατά της ενδυνάμωσης ε, των ανθρώπων ώστε να αποκτήσουν, ε, να ιδιοποιηθούν τη διαδικασία αυτή. Τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν για την καλύτερη παρακολούθηση και τη βελτίωση των πολιτικών μας. Thank you. Uh, next question. Ευχαριστώ πολύ. Από το Renew, κυρία Ροντρίγκε Ράμος. Χωρίς μικρόφωνο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και εγώ για την παρέμβασή σας. Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι μιλάμε για το θεματολόγιο των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης που είναι φιλόδοξο με αλλαγή εστίασης, είναι σαφές αυτό. Και νομίζω ότι η Κομισιόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση εν γέννη θα πρέπει να έχει ηγετική στάση και μέχρι το τέλος ε, να είμαστε πρωτοπόροι και να είμαστε σε θέση να έχουμε ένα θεματολόγιο σαφές με δείκτες ε, και τιμές ενδεικτικές που μέχρι το 2030 θα επιτρέψουν ε, και τις μελέτες αντικτύπου ώστε πριν φτάσει αυτή η ημερομηνία μέχρι τότε να δούμε πώς πρέπει να προσανατολίσουμε τις ήδη φυστάμενε πολιτικές, τι νέες πολιτικές πρέπει να εφαρμόσουμε και πώς πρέπει να χαραχθεί ο προπολογισμό ή να επαναπροσανατολιστεί. Θέλουμε λοιπόν ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση να ηγείται τις προσπάθειες αυτής, άρα πρέπει να ηγειται τις προσπαθειες αυτή, αρα πρεπει να αυξηθει ο προπολογισμό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το είδαμε στον τομέα του περιβάλλοντο. Θέλουμε 25% παραπάνω κονδύλια. Επίσης πρέπει να ηγηθούμε και σε ό,τι αφορά τις αναψώμενες χώρες ώστε να υπάρξει κινητοποίηση πόρων. Αν δεν κινητοποιήσουμε περισσότερους πόρους, οι αναψώμενες χώρες δεν θα μπορέσουν να πετύχουν τους στόχους μέχρι το τέλος αυτής της περίοδου. Εξού και θεωρώ ότι η ευρωπαϊκή ηγεσία πρέπει να δειχθεί, να καταδειχθεί και στο πεδίο της κινητοποίησης εσωτερικών πόρων, δηλαδή στις χώρες με τις οποίες συνεργαζόμαστε. Τους από τους πρασίνους. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Όπως και με τους κλιματικούς στόχους, η έκθεση που μας παρουσιάσατε δείχνει ότι δεν θα πετύχουμε τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης και αυτά τα δύο είναι συνδεδεμένα μεταξύ του θέματα, διότι αυτό που παρατηρούμε όλο και περισσότερο είναι η υποβάθμιση του περιβάλλοντο να πλήττει κυρίω αυτού που βρίσκονται σε πιο ευάλωτη θέση, σε πιο επισφαλή θέση. Μοζαμβίκη, για παράδειγμα, με εκατομμύρια θύματα. Τρία δι δολάρια ήταν οι ζημιέ. Μια σταγόνα νερό στον ωκεανό ε, της υποβάθμισης του περιβάλλοντος, για την οποία είμαστε υπεύθυνοι σήμερα δεν ε, φέρουμε σε πέρα υποχρεώσει μα στον τομέα του περιβάλλοντο και του κλίματο. Το είπατε και εσεί. Θέλουμε παραπάνω χρηματοδότηση. Απαιτούνται περαιτέρω κονδύλια. Πού θα προέλθουν αυτά, από τα κράτη. Αλλά ίσω και με την, ε, την εφαρμογή τη αρχή οριπένων πληρώνει. Έχουμε 25 εταιρείε παγκοσμίω που από το 1998 έως το 2015 ευθύνονται για το 75% των περιβαλλοντικών ζημιών. Αλλά ε, ούτε πληρώνουν επαρκώς και σίγουρα ε, αυξάνονται τα έξοδα ε, για τον κοινό κορβανά από την υπερθέμαση του πλανήτη και άλλες φυσικές καταστροφές. θα έπρεπε ίσως να έχουμε υπόψη ότι υπάρχουν όρια στον πλανήτη. Δεν είναι άπειρο, άπειροι πόροι. Χρειάζονται επίσης και οικονομικοί πόροι ε, και πρέπει να αλλάξουν ε, και οι όροι στήριξης των αναπτυσσόμενων και νομική και οικονομική κλπ. ID, Γκρισέ από ID. Όχι. Όχι. Καλώς. Προχωρούμε τότε. Κέμκα. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Επίτροπε, μας μιλήσατε για τους ε, στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Πάρα πολύ σημαντικό. 169 καθήκοντα στο πλαίσιο 14 στόχων. Τα εθνικά κοινοβόλια, οι τοπικές περιφερειακές αρχές και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συνεργαστούν γιατί χρειάζεται μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, πολυτομεακή προσέγγιση και διαχείριση. Και η κοινωνία των πολιτών θα πρέπει να συνεργαστεί, όπως βέβαια και ο ιδιωτικός τομέας. Άρα Πρέπει να υπάρχει και ιδέωσα παρακολούθηση, να ε, παρακολουθείτε η πρόοδος. Ε, αυτό είναι πάρα πολύ απαραίτητο για τη βελτίωση των εθνικών στρατηγικών σε όλα τα επίπεδα. Και έρχομαι στην ερώτησή μου. Η Μελλοντική Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μιλήσει για τα κενά που υπάρχουν στην στρατηγική αυτή. Θα εντοπίσει τις ε, ανεπάρκειες και τις ασυνέπειες σε ό,τι αφορά στρατηγική μέχρι το 2030. Γιατί έχουμε και το θέμα των στατιστικών, της συλλογής ε, δεδομένων. Γιατί χρειάζεται μία στρατηγική, πλήρη, διεξοδική, ώστε να έχουμε πετύχει τους στόχους του θεματολογίου 2030 ε, και να έχουν κλείσει οι στόχοι αυτοί μέχρι το 2019. Μην ανησυχείτε, είστε όλοι στον κατάλογο των ομιλητών, αλλά προσπαθώ να δίνω το λόγο ε, με τη σειρά λίγο, ανάλογα με το μέγεθος της ομάδας, οπότε μην αρχίσετε να ανησυχείτε αν δεν σας δώσω αμέσως το λόγο. Τώρα και στο όνομα της ΓΚΟΥ, ο κύριος Σπικάρης. Ευχαριστώ. Κόκαλη, συγγνώμη, συγχωρείτε. Η σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να μπορέσουν η Ευρωπαϊκή Ένωση να δείξει παγκόσμια ηγετική ικανότητα και οι στόχοι της, ε, της χιλιατίας είναι αδιαχώρηση από τη Συμφωνία του Παρισιού. Ε, πρέπει να γίνει η μετάβαση στην οικονομία γι' αυτό. Θα πρέπει να μας πείτε πότε και πώς θα εφαρμόσετε το ψήφισμα του Μαρτίου 2019 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έτσι ώστε ο γνώμονάς μας να είναι η στόχη της χιλιετίας και επίσης πώς θα χρησιμοποιηθούν από τη Eurostat ως δείκτες ε, ή στόχοι για το επόμενο PDP. Εάν θέλουμε να επιτύχουμε αυτούς τους στόχους και να περιορίσουμε τις εκπομπές μας, θα πρέπει να θεσπίσουμε ένα νέο ταμείο για την κλιματική μετάβαση τα επόμενα χρόνια. Ευχαριστώ. Η κυρία Ενσύρ. So, now, thank you so much, Chair, and thank you, Commissioner Mimicha, for being here. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, και ευχαριστώ, Επίτροπε Μίμητσα, που είστε εδώ για να συζητήσουμε την ατζέντα για το 2030. Είναι η πρώτη μας ε, συνεδρίαση, είναι και πολύ θετικό που ξεκινάμε με τη συζήτηση ενός τόσο σημαντικού θέματος. Επίσης είπατε κι εσείς ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να παίξει πρωτοποριακό ε, ρόλο για την εφαρμογή των ε, στόχων της χιλιετίας αλλά και τη συμφωνίας του Παρισιού τόσο εντός Ένωσης αλλά και όσον αφορά τις εξωτερικές μας πολιτικές. Πριν να έχω την τιμή να γίνω Ευρωβουλευτής δούλευα με μια ε, μάλλον για τη διεθνή ανάπτυξη μεταξύ άλλων. Από την εμπειρία μου επιτόπου ε, ε, μπορώ να σας πω ότι συχνά υπάρχουν παράλληλες διαδικασίες με ίδιους στόχους αλλά χωρίς συντονισμό από πλευράς δηλαδή Ένωσης και κρατών μελών. Γι' αυτό καταρχάς διερωτάμε, αν μπορείτε κάπως να επεκταθείτε στο θέμα των κοινών προσπαθειών και πώς αυτές μπορούν να αναπτυχθούν. Έπειτα θα ήθελα να ξέρω πώς βλέπετε το δυνατότητα να αναπτυχθούν προσεγγίσεις όπως για παράδειγμα η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι καλύτερη στην πρόθεση της ισότητας των φύλων και σίγουρα σε σχέση με τη διάσκεψη κορυφής του Σεπτεμβρίου. Και με ποιους τρόπους η Ευρωπαϊκή Ένωση θα γίνει καλύτερη ε, στην προώθηση του κοινωνικού διαλόγου ως ε, μέσου για τη μείωση των ανισοτήτων ανάμεσα στους ε, ε, λαούς και στις περιφέρειες. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γκέρνς είναι ο τελευταίος για αυτό το γύρο ερωτήσεων. Μάλιστα σας ευχαριστώ. Η ερώτησή μου είναι απλή. Η Κομισιόν έχει μία εκ των ε, προτέρων αξιολόγηση για τον αντίκτυπο που θα έχει η Συμφωνία Μερκοσούρ που μόλις τελείωσαν οι διαπραγματεύσεις ε, για αυτήν όσον αφορά τους στόχους για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Πολύ σύντομη και περιεκτική ερώτηση σας. Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, μπορείτε να απαντήσετε στις ερωτήσεις εξίσου συντόμως και περιεκτικά. Θα το εκτιμούσαμε όλος ιδιαίτερος. Σας ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις σας και τα σχόλιά σας και για τις συμβολές, τη συμβολή σας στη δουλειά, στο έργο που έχουμε ενώπιόν μας να καταστήσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση τον βασικό μέτοχο στην εφαρμογή των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης. Υπήρξαν πιο συγκεκριμένες και πιο γενικής φύσης ερωτήσεις. Θα προσπαθήσω να απαντήσω κάπου πρώτα σε πιο συγκεκριμένες ερωτήσεις για την εφαρμογή των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης για την ε, υγεία. Η δική μας συμβολή στην ε, ανθρώπινη ανάπτυξη μέσω, όσον αφορά δηλαδή την υγεία, την παιδεία, όλα αυτά εντάσσονται στο πλαίσιο των εθνικών μας ε, δικτικών προγραμμάτων και φακέλων, αναπτυξιακών φακέλων, όπου εργαζόμαστε εντόνως και θα θέλαμε να αυξηθεί η δέσμευση όσον αφορά τη βελτίωση των συστημάτων υγείας σε επίπεδο χωρών και ο δεύτερος άξονας είναι η οικονομική στήριξη αλλά και η στήριξη μέσω πολιτικών των κάθε των παγκόσμιων πρωτοβουλειών όπως το Παγκόσμιο Ταμείο για την καταπολέμηση της ελονοσίας, της φυματίωσης του AIDS ή οργανισμών όπως αυτός του Μουγκάμπε. Επίσης να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τα συστήματα υγείας να ανταποκριθούν στις ε, ανάγκες υγείας και να οδηγηθούμε σε αριστεία ώστε να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη του ανθρωπίνου κεφαλαίου, στην ανάπτυξη των συστημάτων υγείας στην επόμενη περίοδο. Όσον αφορά την ανισότητα, φυσικά συμφωνώ ότι πρόκειται για ένα θέμα που διέπει όλα τα υπόλοιπα που μπορεί να αποτελέσει την κινητήριο δύναμη για όλα τα υπόλοιπα θέματα ή και να μειώσει το θετικό αντίκτυπο που μπορεί να έχει αναπτυξιακή συνεργασία σε ε, για την επίτευξη των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης. Σίγουρα λοιπόν στο μέλλον θα πρέπει να εστιάσουμε περισσότερο την προσοχή μας και να είμαστε πιο συγκεκριμένοι όσον αφορά τις δράσεις μας σχετικά με τις ανισότητες. Έχουμε έναν γενικό στόχο που προκύπτει από την Παγκόσμια Ατζέντα για τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης Εάν λοιπόν συνδυάσουμε το ότι δεν θέλουμε κανέναν να αφήσουμε εκτός και τις πολιτικές μας περιμείωσης των ανισοτήτων, πιστεύω πως θα δώσουμε μεγαλύτερη όθηση στην επίτευξη των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης. Ε, βέβαια, ίσως ε, είναι κάπως αργά για να σας δώσω ένα γενικό πλαίσιο για έναν επίτροπο που θα φύγει σε τρεις μήνες, αλλά οι πολιτικές μας θα πρέπει να αναπτυχθούν προς μια κατεύθυνση έτσι ώστε να φτάσουμε σε ένα επίπεδο όπου να έχουμε δείκτες νησοτήτων, όπως έχουμε τους, ε, ε, για τις δράσεις που σχετίζονται με το φύλλο, ώστε να μπορούμε εύκολα να εκτιμήσουμε να και να παρακολουθήσουμε πώς συμβάλλει κάθε αναπτυξιακό πρόγραμμα στην μείωση των ανισοτήτων. στις χώρες εταίρους μας. Το έχουμε για τις δράσεις για το φύλλο. Υπήρξε και ένα ερώτημα για το πώς μπορούμε να καταστήσουμε τη δράση μας για το φύλλο πιο αποδοτική, αποδοτικές και θα ήθελα να σας πω ότι μέσα στο πρόγραμμά μας ε, δράσεις έχουμε τοποθετήσει ένα σαφή στόχο ότι τουλάχιστον 85% όλων μας των αναπτυξιακών προγραμμάτων θα πρέπει να έχουν σχέση με το φύλλο. Τώρα ε, κοντεύουμε στο 70% των αναπτυξιακών μας δράσεων και θα θέλαμε το ίδιο να γίνει και στον τομέα της ισότητας. Εν γέννη, η παρακολούθηση και η βελτίωση της λογοδεσίας σε σχέση με τις αναπτυξιακές μας δράσεις είναι ένα σημαντικό ε, κομμάτι της εφαρμογής των, ε, των δράσεων βιώσιμης ανάπτυξης. Πρέπει να στραφούμε από το input στο output. Να μετράμε και να εστιάσουμε στο ποιο είναι το αποτέλεσμα των αναπτυξιακών μας ε, προγραμμάτων. Γι' αυτό και τα αποτελέσματα της αναπτυξιακής μας συνεργασίας θα είναι ένα πολύ σημαντικό τμήμα της αναπτυξιακής μας πολιτικής και η δική μας συμβολή στην εφαρμογή των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης. Για την Ευρωπαϊκή Ένωση είμαι βέβαιος ότι θα συνεχίσουμε να είμαστε ο ισχυρότερος παγκόσμιος φορέας στις αναπτυξιακές πολιτικές και αυτό ε, ελπίζω πως θα αντικατοπτριστεί και με τη δική σας αναγνώριση, κατανόηση και συμβολή αυτό θα αντικατοπτρίζεται και στο επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Διότι αυτό που έχει, που έχει προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι μια αύξηση περίπου 30% για όλες τις εξωτερικές δράσεις και για την αναπτυξιακή συνεργασία. Να έχουμε δηλαδή περισσότερες δυνατότητες να είμαστε παγκόσμιος ε, ηγέτης στην αναπτυξιακή χρηματοδότηση συμβαδίζει με την ευθύνη που φέρουμε για την εξέβρεση του καλύτερου τρόπου για την λογοδοσία των αναπτυξιακών μας ε, δράσεων βεβαίως. Κάποιες φορές και μπορεί να υπάρχουν και υπάρχουν και να οι επικαλύψεις στις στρατηγικές μας, ιδιαίτερα αν έχουμε υπόψη μας <coughs> ότι έχουμε 28 μέλη και διάφορα ευρωπαϊκά μέσα που συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη και στην εφαρμογή των σχετικών στόχων. Γι' αυτό Ήδη ε, ξεκινήσαμε στη διάρκεια του τρέχοντος PDP, ξεκινήσαμε με ένα καλύτερο πρόγραμμα, με μια προσπάθεια μάλλον καλύτερου προγραμματισμού, έτσι ώστε τα κράτη-μέλη μας, αλλά και κάποιες από τις τρίτες χώρες, όπως η Αυστραλία, η Αυστραλία, ο Καναδάς, η Ιαπωνία, η να είμαστε πιο συντονισμένοι. Στο μέλλον λοιπόν η εφαρμογή των αναπτυξιακών στόχων μέσω αυτών των κοινών προγραμμάτων θα είναι πιο ε, σημαντική. Τώρα για τη συσχέτιση μεταξύ της Συμφωνίας του Παρισιού και των ε, στόχων βιώσιμη ανάπτυξη αλλά και τη κλιματική δράση, δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα περισσότερο παρά να τονίσουμε το γεγονό ότι η, η έννοια ε, των στόχων βιώσιμη ανάπτυξης είναι ακριβώς η βιωσιμότητα, η συμπερίληψη κλιματικών προβληματισμών και δράσεων στην αναπτυξιακή δράση. Και αυτό ακριβώς και θα κάνουμε ε, με βάση τη συνένεση για την ανάπτυξη που θα μπορούσε ίσως κανείς να το δει ως τη δική μας στρατηγική για την εφαρμογή των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης. Αλλά κατανοώ απόλυτα την έκκληση του Κοινοβουλίου και της κοινωνίας των πολιτών η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναπτύξει ακόμα πιο συγκεκριμένη και λεπτομερή στρατηγική για την εφαρμογή των αναπτυξιακών στόχων μέσω της Ευρωπαϊκής Συνένεσης για την Ανάπτυξη. Βλέπω δηλαδή ότι αυτή θα πρέπει να είναι η κατεύθυνση που θα πρέπει να ακολουθήσει η επόμενη Επιτροπή. Ελπίζω έτσι να, να, απάντησα για το Μερκοσούρ. Τελευταίο λεπτό που σας δίνουμε. Όπως σε όλες μας τις συμφωνίες και τις διαπραγματεύσεις μάλλον για τις ε, συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου ε, προβαίνουμε σε εκτίμηση αντικτύπου εξάντε εκ των προτέρων. αυτό έχει γίνει και για την Συμφωνία εμπορίου με τις χώρες του Μερκοσούρ. Έχουν γίνει μάλιστα δύο τέτοιες αξιολογήσεις, μια εσωτερική και μια εξωτερική. Και οι δύο δείχνουν τα κέρδη και για τη βιώσιμη ανάπτυξη που θα προκύψουν από αυτήν την μεγάλη εμπορική συμφωνία ελευθερού εμπορίου που έχουμε ποτέ συνάψει, η οποία δεν είναι μόνο μεγάλη λόγω του όγκου του εμπορίου που καλύπτει, αλλά είναι και μεγάλη όσον αφορά τα καινοτόμα τμήματα της συμφωνίας και τις προδιαγραφές που καλύπτονται από τη Συμφωνία Μερκοσούρ. Thank you. Σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Θα συνεχίσουμε, θα ακούσουμε και άλλες ερωτήσεις από τους Ευρωβουλευτές, ε, από το ΕΛΚ ή η Μαρή Μακίνες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ συνάδελφοι. Μία παρατήρηση. Χαίρομαι που μας θυμήσατε ότι οι στόχοι αυτοί ε, αναφέρονται και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ε, μας ενδιαφέρει μόνο η εξαγωγή τους. Ε, δεύτερον, βιώσιμη γεωργία, επιστημιστική ασφάλεια και διατροφή. Η σχετική έκθεση είναι αρκετά απεσιόδοξη λόγω της έλλειψης πρόοδου στα θέματα αυτά. Ένα από τα θέματα που τονίζονται στην έκθεση είναι ότι υπάρχει μείωση δημοσίων επενδύσεων στη Γεωργία και αναρωτιέμαι, η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει αρκετά στον αναπτυσσόμενο κόσμο για να στηρίξει τη Γεωργία διότι αναφέρονται τα προβλήματα ε, των ε, γεωργών μικρής κλίμακες ε, και η μεταφορά τεχνογνωσίας ε, είναι όντως κατάλληλη για τις περιφέρειες αυτές. Κάνουμε αρκετά σε αυτές τις περιφέρειες. Η έκθεση είναι πολύ απεσιόδοξη στο θέμα αυτό. Απογοητευτικό τέσσερα χρόνια μετά. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Μόνικα Κονσάλης από το S&D. μικρόφωνο. Συγγνώμη, συγγνώμη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Εγώ ε, θεωρώ ότι είναι πολύ συναρπαστικό αυτό που συζητάμε σήμερα, το θέμα του 2030 και η στόχη βιώσιμη ανάπτυξη. Από το 2014 σήμερα κάνετε σημαντική προσπάθεια, μεταξύ άλλων το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Επενδύσεων με την Αφρική, 44 εκατομμύρια ευρώ, ούτε λίγο ούτε πολύ. Βέβαια, άργησε η Κομισιόν να ενσωματώσει τους στόχου βιώσιμη ανάπτυξη από ό,τι καταλαβαίνω στο θεματολόγιο τη ε, Κομισιόν εν γέννη. Συμφωνώ ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να διατυπώσει πιο συγκεκριμένε προτάσει ενδεχομένω από αυτέ που περιλαμβάνει η συναντική πρόταση του 2017 μεταξύ Συμβουλίου Κοινοβουλίου και Κομισιόν. Πιστεύω ότι πράγματι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ηγηθεί απέναντι σε αυτή την επίθεση σε βάρο του πολυμερού συστήματο, όπω βλέπουμε από τη Ρωσία, από τη ΣΥΠΑ. Πρέπει λοιπόν να είναι ηγετική η θέση σε τρία θέματα. Το πρώτο είναι η μείωση των ανισοτήτων η ισότητα των δύο φίλων πάρα πολύ σημαντική για τη βιώσιμη ανάπτυξη και είναι στον πυρήνα των αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι πρωτοβουλίε ε, των οποίων γεθήκατε εσεί είναι σημαντικέ, αλλά υπάρχουν οι ε, άνθρωποι και πρέπει νομίζω να περιλάβουμε ε, την πολυμορφία, του σελοάδμα, την αναπηρία και δεύτερο, εγκάσιο χαρακτήρα. Είναι πολύ σημαντικό νομίζω να δημιουργηθούν συμμαχίες ε, και μέτωπα με ΜΚΟ, τοπικούς φορείς, δήμους, ε, ε, περιφερειακές τοπικές αρχές. Και τρίτον, δίκαιη μετάβαση, ακριβώς για να ενισχύσουμε οικολογική μετάβαση για τις πιο ευάλωτες περιοχές του κόσμου, η Λατινική Αμερική, η Αφρική. Η, Ήπουρο, που δεν ευθύνεται, ευθύνεται το λιγότερο για τις εκπομπές, αλλά πλήττεται περισσότερο από την κλιματική αλλαγή πέρυσι και ήταν σημαντικό αυτό που έγινε, εγκρίναμε το Παγκόσμιο Σύμφωνο για τους πρόσφυγες. ενέργεια και Γκερέρο ήταν ο σύντροφό μας που πολλές φορές πρότασε, ε, πρότεινε να υπάρξει η έννοια του κλιματικού πρόσφυγα. Πριν λήξει η θητεία σας, ε, θα ήταν καλό να έχετε μια συγκεκριμένη πρόταση για να δοθεί ε, ένα προφίλ σε αυτού του είδους τους πρόσφυγες να ρυθμιστούν αυτά, πιστεύω, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό στο πλαίσιο της θείας. Σας ευχαριστώ. Thank you. Uh, we try to keep... Σας ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ ε, να προσπαθείτε να περιοριστείτε στο ένα λεπτό. Renew Europe. Excusez-moi, je sais pas. Euh, bon, bonjour, merci, euh, commissaire. Ε, okay, uh, σας ευχαριστώ Επίτροπε και ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι για αυτή τη συνεδρίαση γιατί εγώ είμαι μέλος και των δύο επιτροπών της ε, ανάπτυξης και του περιβάλλοντος. Εγώ έχω μια γενική φύση ερώτηση. Είμαι νεοεκλογή σας στο Ευρωκοινοβούλιο. Και Χαίρομαι για τη μεγάλη φιλοδοξία που δείχνει η Κομισιόν, αλλά διαρωτώ με πώς να μην γίνει κανείς χιζοφρενής, πώς να μην ε, φτάσει να κάνει ε, πραγματικά τους στόχους ε, της βιώσιμης ανάπτυξης αλλά και τους, της Συμφωνίας του Παρισιού κάτι που να είναι ε, να διέπουν όλους τις πολιτικές της Κομισιόν δηλαδή να είμαστε πραγματικά συντονισμένοι σε όλες τις εργασίες που μας περιμένουν πάνω σε αυτούς τους στόχους. Ευχαριστώ. Από το ECR η κυρία Σελεύσκα. Panie komisarzu, stwierdził pan, że... Σας ευχαριστώ πολύ. Είπατε ότι ως Ευρωπαϊκή Ένωση θέλουμε να είμαστε οι πρώτοι όσον αφορά την ε, προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης σε όλο τον κόσμο. Ε, συμφωνώ, για να είμαστε καλύτεροι όμως πρέπει να δώσουμε καλά παραδείγματα και χρειαζόμαστε έτσι καλή ισορροπία ανάμεσα στα ωφέλη ε, και τις απώλειες. Και επίσης θα πρέπει να προγραμματίσουμε σωστά αυτά που θέλουμε να κάνουμε στο μέλλον. Κύριε Επίτροπε, και επίσης ε, συμμετείχατε στις διαπραγματεύσεις ε, για το προσεχές πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Τι προτάθηκε λοιπόν εκεί. Εγώ πιστεύω ότι πολλές προτεραιότητες αποκλείουν η μία την άλλη. Αν σκεφτόμαστε την γεωργία, δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να μειωθεί το εισόδημα των ε, γεωργών. Ε, χρειάζονται χρήματα για να προστατευτεί το έδαφος. Σας παρακαλώ λοιπόν να απαντήσετε στην ερώτησή μου. Σας ευχαριστώ. Δόμινικ Πίλτα από την IND. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε για τις εξηγήσεις που μας δώσατε για τους στόχους της ευγιώσιμης ανάπτυξης. Ε, πώς θα συμπεριληφθούν στο ευρωπαϊκό εξάμεινο. Αυτό είναι το πιο δύσκολο. Δεν θα είχαν αυτονομία τα κράτη-μέλη, όπως σε θέματα ενεργειακά, όπου η Ένωση ανεπιφύλακτα στηρίζει τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αν και γνωρίζουμε πόσο προβλήματα δημιουργούν οι ανεμογεννήτριες. Έχουμε και την έκθεση Eurostat, που φαίνεται να κρύβεται ο διάβολος στις λεπτομέρειες. Είναι ενδιαφέρον λοιπόν να διαπιστωθεί ότι αυτή η έκθεση ουσιαστικά ως θετικό παρουσιάζει την αύξηση των εμπορικών συναλλαγών με τι ανεψόμενε χώρες. Περιλαμβάνει και την Κίνα όμως. Ενώ η Κίνα κάνει μαζικό dumping σε βάρος των δικών μα βιομηχανιών. Σε ό,τι διαφορά εισαγωγέ από λιγότερο προηγμένε, όπως λέγονται, χώρες, που μεταξύ τους είναι και κάποιε γαλλόφωνε. 2% μόλις είναι σε αυτές τις συναλλαγές. Στην έκθεση επίση λέγεται ότι είμαστε ήδη ε, σε μια εποχή που η Κίνα ελέγχει μεγάλο μέρος της Αφρικανικής Υπήρου και ξεπερνάει την Ένωση. Πώς θα μειωθεί η εξάρτησή μας απέναντι στην Κίνα πώς θα πάψουμε να κρατήσει για τον εαυτό της και ως ε, λάφυρο την Αφρικανική Υπήρου. Ευχαριστώ. S&D Roy Palmer. Σας ευχαριστώ. Αύριο, τέτοια ώρα, ένα από τα κράτη-μέλη μας θα έχει νέο πρωθυπουργό. Νέο πρωθυπουργό που είπε ότι θέλει να κλείσει το ε, Υπουργείο ε, Διεθνούς Βοήθειας ε, του Ηνωμένου Βασιλείου, που θέλει να ευθυγραμμίσει την αναπτυξιακή βοήθεια του Ηνωμένου Βασιλείου για να στηρίξει ε, εμπορικά, οικονομικά συμφέροντα. Και νομίζω ότι είναι σημαντική αυτή η στιγμή για τους ανθρώπους που θέλουν πολυμερή προσέγγιση. Θα πρέπει να δούμε αποτελέσματα όσον αφορά τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Εάν λοιπόν έχετε ένα μήνυμα για τον ε, μελλοντικό πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον, τι θα ήταν αυτό το μήνυμα. Ευχαριστώ από τη Renew Europe, ε, Μάρτιν Χολ. Σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε, πολύ χαίρομαι που μιλήσατε για την παρακολούθηση, θέμα κάπως βαρετό, αλλά πάρα πολύ σημαντικό, ε, εάν θέλουμε το πολιτικό φόρουμ υψηλού επίπεδου να ε, διαπιστώσει ε, εάν ε, πετυχαίνονται οι στόχοι και οι 230 δείκτες που τους στηρίζουν. Σε όλο τον κόσμο οι φτωχότεροι αποκλείονται από τα επίσημα δεδομένα και αν κοιτάξετε το φτωχότερο 20%, σχεδόν το μισό των παιδιών κάτω των 5 ετών δεν έχουν καν ε, καταγραφεί στο ληξιαρχείο. Δηλαδή δεν έχει καταγραφεί η γέννησή τους ε, και έτσι δεν έχουν πρόσβαση στην υγεία, ε, δεν έχουν άλλα δικαιώματα και έτσι ποτέ δεν γνωρίζουμε αν οι φτωχότεροι έχουν ξεχαστεί ή όχι. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι... Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα επενδύσει στα ληξιαρχικά συστήματα, στα συστήματα διοικητικών δεδομένων, ώστε να διασφαλίσουμε ότι οι φτωχότεροι δεν είναι αόρατοι σε όλη αυτή τη διαδικασία. Ευχαριστώ και η Ελεονόρα Εύη. Τελευταία ερώτηση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εδώ βρίσκομαι, Επίτροπε. Καταρχάς, ευχαριστώ για την εργασία σας στη διάρκεια της θητείας σας. Εγώ επανέρχομαι σε μια ερώτηση που υπέβαλαν ήδη συνάδελφο και που έχει αποτελέσει αντικείμενο ψηφίσματος του Ευρωκοινοβουλίου στην περασμένη θητεία και που αφορά ακριβώς την γενική, τη σφαιρική στρατηγική για ενημέρωση της Ατζέντα 2020 που περιλαμβάνει μέτρα και συγκεκριμένα ε, και στόχους με συγκεκριμένες προθεσμίες. Οπότε πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος μέτρησης ε, για την κατάσταση πρόοδου. Και αυτό το είχε ζητήσει από την προηγούμενη θητεία το Ευρωκοινοβούλιο. Εσείς σήμερα το αναφέρατε, αλλά πιστεύω πως είναι αυτή εδώ στιγμή πολύ σημαντική και χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση να στήσει και αυτή τη γενική σφαιρική στρατηγική. Και επειδή το είπε και η συνάδελφος που μίλησε πριν από μένα, για παράδειγμα για τα παιδιά. Τα παιδιά είναι ζουν σε δραματικές συνθήκες ε, πολλές φορές εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκτός ε, των συνόρων της Ένωσης. 37 είναι τα κράτη τα οποία δεν έκαναν επαρκή πρόοδο σε σχέση με τις ε, στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης όπως λέει η UNICEF και μισό, εκατομμύριο, μισό δισεκατομμύριο είναι ε, τα παιδιά που ζουν σε χώρες όπου δεν έχει γίνει καμία απολύτως πρόοδο. Τι σκοπεύετε να κάνετε σε σχέση με αυτό το σημαντικό θέμα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και σας ευχαριστώ όλους συνάδελφοι για τις ερωτήσεις. Δίνω το λόγο στον Επίτροπο και πάλι. Yes, on... Σας ευχαριστώ. Πράγματι, εδώ και δεκαετίες η πείνα στον κόσμο μειώνεται. Δυστυχώς όμως, από το 2015, όπως λέει ΦΑΟ, βλέπουμε να αυξάνεται το φαινόμενο. Παρά των πραγματικά μεγάλων προσπαθειών που καταβαλώ όχι μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά η διεθνής κοινότητα εν γέννη. Για να εστιάσει σε θέματα ασφάλειας τροφίμων και διατροφής εν γέννη. Στο πλαίσιο του ΠΔΕΛΤΑΠΗ που ισχύει, δεσμεύσαμε σχεδόν 8 και πάνω ε, δις σε προγράμματα που σχετίζονται με τα τρόφιμα και σκοπεύουμε να συνεχίσουμε στην ίδια κατεύθυνση πιο συγκεντρωμένα, πιο εστιασμένα και ισχυρά με τους εταίρους μας, ΦΑΟ και λοιπούς. Φορείς και κρατημέλη και άλλους stakeholders. με την ε, αύξηση κατά 30% σχεδόν σε όλες αυτές τις εξωτερικές δράσεις θα μπορούσαμε να έχουμε περισσότερες δράσεις ε, και να χρηματοδοτήσουμε καλύτερα τα προγράμματα που σχετίζονται με τα τρόφιμα. Σίγουρα λοιπόν τρόφιμα γεωργία παραμένουν ψηλά στις προτεραιότητες. Και σε ό,τι αφορά τις παρεμβάσεις ε, από την αναπτυξιακή πολιτική για την επιτευχή στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης. Πολλές φορές ακούστε και από εσάς η ανάγκη μεγαλύτερης διασύνδεσης ε, της δράσης για την κλιματική αλλαγή και της αναπτυξιακής δράσης. Θέλω να επιστήσω την προσοχή σας στο γεγονός πως όπως ήδη προανέφερα, αυτό που κάνουμε τώρα και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε, είναι ότι συνεργαζόμαστε με τα κράτη-μέλη για την κατάρτιση των εθνικών ε, αναπτυξιακών τους σχεδίων, ολοκληρωμένα σχέδια αυτά. Αλλά δεν το βλέπουμε απομονωμένα σε σχέση με άλλες πολιτικές. Γιατί πρέπει να υπάρχει μία συνεκτικότητα. Άρα θα επιμείνουμε ώστε οι εθνικές ανεπεξίες στρατηγικές των χωρών εταίρων να συνδυαστούν με τις εθνικά καθορισμένες συνεισφορές, τα NDCs, σε σχέση με την κλιματική αλλαγή. Για μας πρόκειται για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση. Δηλαδή αναπτυξιακές δεσμεύσεις και κλιματικές δεσμεύσεις από κοινού. Θα αυξήσουμε γενικά την αναπτυξιακή υποστήριξη και ενίσχυση που παρέχουμε στους αναπτυξιακούς μας εταίρους. Ο στόχος που προτείνουμε είναι 25% του συνόλου των αναπτυξιακών δράσεων ώστε να έχουν σχέση με το κλίμα. Βέβαια αυτό εξαρτάται από το Κοινοβούλιο, από τα κράτη-μέλη και από την Κομισιόν εν γέννη, για να καθορίσει ένα οριστικό επίπεδο. Μπορεί το 25% να είναι χαμηλό ή ψηλό, δεν ξέρω, δεν μπορώ να πω εγώ. Είναι αυτός πάντως ένας τομέας ακόμη που το σκέλος της ανάπτυξης ε, θα, θα πρέπει να συνδυαστεί με το σκέλος του κλίματος. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ακούστε, Σίγουρα πρέπει να παραμείνουμε προσιλωμένοι στην στήριξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την ανάπτυξή τους στον κόσμο ολόκληρο. Η αναπτυξιακή συνεργασία και τα σχετικά της προγράμματα. Δεν θα πρέπει να χρηματοδοτεί οποιαδήποτε άλλη μορφή για την παραγωγή ενέργειας ε, ηλεκτρικής πλήν ε, ε, των ανανεώσιμων. 40 εκατομμύρια άνθρωποι θέλουμε να έχουν πρόσβαση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Τουλάχιστον 40 εκατομμύρια. 6,5 γιγαβάτ ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Άλλος ένας στόχος. Άλλος στόχος. 15 εκατομμύρια τόνοι εκπομπών του άνθρακα να έχουν ε, πάψει να εκλείονται μέχρι το τέλος του 2020. Με όλους αυτούς τους στόχους για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας νομίζω ότι παραμένουν προσιλωμένοι στην αναπτυξιακή μας πολιτική και αποφασιστική. Συμφωνώ ότι μπορεί να υπάρχει κάποιος διαβολάκος που να κρύβεται στις λεπτομέρειες, αλλά εμείς θα τον βγάλουμε από όπου και αν κρύβεται και δεν υπάρχει κρυφές ατζέντε για τις βιώσιμες πηγές ενέργειας. Θα παραμείνει στον πυρήνα των δράσεών μας τώρα. Να σας πω έτσι σύντομα δύο πράγματα σε ό,τι αφορά την Κίνα. <clears throat> Δεν θα ήθελα να υποβαθμίσω το ρόλο της Κίνας στην αναπτυξή πολιτική, ιδίως στην Αφρική. Όμως, μέχρι στιγμής, η Ευρώπη, τα κράτη-μέλη, η Ευρωπαϊκή Ένωση, μακράν είναι ο μεγαλύτερος αναπτυξιακός εταίρος της Αφρικής, ο μεγαλύτερος επενδυτικός εταίρος και ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Αφρικής. 40% άμεσων ξένων επενδύσεων πάνε στην ε, Αφρική, η Κίνα είναι στο 5% ακόμη. Άρα με αυτό το φωτογραφικό στιγμιότυπο αν θέλετε δεν σημαίνει ότι θεωρούμε ότι είμαστε και καλύτεροι και δεν πρέπει να αλλάξει τίποτα, αλλά απλά για να βάλω τα πράγματα σε ένα επιπλαίσιο και στο διάλογο που θέλουμε να έχουμε με την Κίνα, ο στόχος μας είναι σε αυτά τα πιλωτικά προγράμματα σε κάποιες χώρες να δούμε κατά πόσο θα ήταν δυνατόν να προωθήσουμε συμπληρωματικά μεταξύ τους αναπτυξιακά προγράμματα, αντί του να υπάρχει μια συγκρουσιακή σχέση, μια αντιπαράθεση μεταξύ των δύο πλευρών σε αυτά τα αναπτυξιακά έργα. Δεν είμαστε ακόμα εκεί. Δεν έχουμε ακόμη συμφωνήσει για τρεις τουλάχιστον πολιτικές χώρες, αλλά έτσι θα θέλαμε. Θα θέλαμε να υπάρχει μεγαλύτερη συμμόρφωση και λιγότερος ανταγωνισμός στις σχέσεις μας και τη συνεργασία μας για τα θέματα τα αναπτυξιακά και ιδίως ό,τι αφορά την Αφρική. Επίσης, η ψηφιακή τεχνολογία την ανάπτυξη ε, προσλαμβάνει όλο και μεγαλύτερη σημασία. Θέλουμε λοιπόν να στηρίξουμε μέσω αυτού και τις αναπτυξιακούς στόχους και έχουμε ένα συμπεφωνημένο πρόγραμμα που αποσκοπεί στη μεγαλύτερη ψηφιοποίηση. Για να υπάρχει καλύτερη κάλυψη των διαφορών στην Αφρική, Δυτική Αφρική. Ενημέρωση και ψηφιοποίηση πολλών μητρών ήδη έχει ξεκινήσει στη Δυτική Αφρική. Και έτσι θα συνεχίσουμε. Αυτή θα είναι μια σημαντική συνεισφορά και δεν μιλώ μόνο για τα μητρώα τα ληξιαρχικά, για τα ληξιαρχεία αλλά και για άλλα. Γιατί όλα αυτά θα βοηθήσουν και τη δημιουργία θέσεων εργασίας ε, στο μέλλον. Perfect. Ε, Τέλεια. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Επίτροπε, που απαντήσατε στις ερωτήσεις των Ευρωβουλευτών. Σημαντικά πράγματα μας περιμένουν. Ο ο Επίτροπος ε, πρέπει να αποχωρήσει. μη φύγετε όλοι, έχουμε κι άλλα. Κύριε Επίτροπε, εμείς εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο θα προετοιμαστούμε, θα σας δούμε στη Νέα Υόρκη για τη συνάντηση κορυφής. Πρέπει και εμείς να βρούμε έναν επικοδομητικό τρόπο να εφαρμόσουμε τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας αφιερώσατε το χρόνο σας. Yes, uh, we also at this uh, meeting. Uh, Έχουμε τη χαρά σήμερα να μπορούμε να ακούσουμε περισσότερες παρατηρήσεις Έχουμε εδώ την ε, Γενική Διευθυνσή για το Κλίμα, έχουμε και εκπρόσωπο της ΕΙΕΔ στη σημερινή συνάντηση. Θα σας δώσω λοιπόν το λόγο για να σχολιάσετε περαιτέρω αυτά που είπε ο Επίτροπος. Πρώτα, δίνω το λόγο στον Ραφαήλ Μωρίς Πεθιόν. Παρακαλώ. Thank you, Chair. Good afternoon. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλό απόγευμα σε όλους. Μία πολύ σύντομη παρατήρηση που σχετίζεται με μία από τις απαντήσεις. Σας παρακαλώ, διακόπτει ο Πρόεδρος. Θέλουμε να ακούσουμε τι έχει να μας πει η Γενική Διευθυνσία για το κλίμα και θέλουμε επίσης να βλέπουμε τον εκπρόσωπό της. Εντάξει, τώρα ρωτάει ο μιλητής. Μία σύντομη παρατήρηση για το πρότυπο ανάπτυξης που προσφέρουμε σε αναπτυσσόμενες χώρες. Νομίζω ότι το πρότυπο μας είναι ουσιαστικά νεκρό. Το παλαιό πρότυπο ήταν ότι βοηθάμε τις αναπτυσσόμενες χώρες να αναπτυχθούν, να γίνουν σαν και εμάς. Αλλά αυτό τελικά έχει αρνητικά αποτελέσματα όσον αφορά το κλίμα. Τώρα λοιπόν αυτό που προσφέρουμε δεν έχει αποδείξει ακόμη την αξία του και αυτό είναι ένα από τα οξύμορα της προσέγγισής μας. Για να ενισχύσουμε την αξιοπιστία του μοντέλου θα πρέπει ε, να ε, αλλάξουμε πρότυπο. Και το παράδειγμα των, βιο... των ε, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι πολύ καλό. Πρέπει να πείσουμε τις αναπτυσσόμενες χώρες ότι πρέπει να επενδύσουν στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και αυτό θα πρέπει να το κάνουμε επειδή το έχουμε κάνει και εμείς και έχουμε αποδείξει ότι λειτουργεί καλά. Αλλά απ' την άλλη θα είναι δύσκολο να πείσουμε 800 εκατομμύρια Αφρικανών που δεν έχουν πρόσβαση σε πηγές ενέργειας να ε, προσπεράσουν τα ορυκτά καύσιμα ε, και να προχωρήσουν στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αν εμείς συνεχίσουμε να καίμε άνθρακα και δεν προχωρήσουμε σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και ξέρουμε ότι το δικό μας πρότυπο ανάπτυξης δεν θα αλλάξει εν μία νυχτή. Έχουμε ένα σχέδιο για να αλλάξει. Τώρα συζητάμε πώς μπορούμε να αναπτύξουμε περαιτέρω το σχέδιό μας. Ε, ούτε προτείνω να μην κάνουμε τίποτα στι αναπτυσσόμενες χώρες μέχρι να συγυρίσουμε το δικό μας νοικοκυριό. Αλλά θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες βλέπουν αυτή την αντίφαση. Σας ευχαριστώ πολύ. Δίνω το λόγο στον κύριο Κριστιαν Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, συνεχίζοντας ε, πάνω σε αυτά που είπε ο Μάριο Πετριτσιόν, ε, με τα οποία συμφωνώ απολύτως, ε, θα ήθελα να αναφερθώ και σε μία παρατήρηση που έγινε πριν. Ήδη ενσωματώνουμε τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης στις πολιτικές μας σε εσωτερικό και εξωτερικό επίπεδο. Εγώ βέβαια κυρίως μπορώ να μιλήσω για την εξωτερική πτυχή. Τα δύο κυριότερα πλαίσια που έχουμε αναπτύξει, το ένα μάλιστα με την υποστήριξη και καθοδήγηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είναι η συνένεση για την ανάπτυξη, που πριν λίγα χρόνια στηρίχθηκε ρητά στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης ως το γενικό πλαίσιο πολιτικής για την μελλοντική αναπτυξιακή μας ε, βοήθεια. Το άλλο είναι η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας. Μπορεί να εκπλήσει με την πρώτη ματιά ότι ένα έγγραφο εξετάζει κυρίως την ασφάλεια των, ε, πολιτικο... των Ευρωπαίων πολιτών, ε, αλλά προσανατολίζεται πολύ ισχυρά στις... Ε, στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Με τη δεύτερη ματιά όμω αυτό δεν εκπλήσει, διότι ε, η ευημερία και η ασφάλεια σε άλλα μέρη του κόσμου αποτελεί την καλύτερη εγγύηση για την ασφάλεια και ευημερία και στην Ευρώπη. Πολύ χαρήκαμε με τη σημερινή κοινή συνάντηση της ΕΝΒΗ και της ΔΕΒΕ. Διότι με πολλούς τρόπους δείχνει το το πρότυπο, το μοντέλο της τούρτας γάμου, όπου βλέπουμε τα διάφορα επίπεδα. Για παράδειγμα, αν δεν φροντίσουμε τους ωκεανούς, όλα τα άλλα θα πάνε χαμένα. Θα πρέπει να φροντίσουμε λοιπόν όλες οι πολιτικές μας, εσωτερικές και εξωτερικές, όσον αφορά τη συνεργασία μας με άλλα μέρη του κόσμου, αναπτυξιακή συνεργασία ή άλλη συνεργασία. Θα πρέπει να φροντίσουμε λοιπόν όλες αυτές οι πολιτικές να στηρίζουν τους στόχους μας όσον αφορά την αλλαγή του κλίματος. Και γι' αυτό στις προτάσεις στο νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο όσον αφορά τις εξωτερικές πιστώσεις τονίζουμε τους κλιματικούς στόχους ως στόχους και για άλλα συστήματα. Και δεν εκπλήσει τα θεσμικά όργανα ότι και το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν δείξει, έχουν δηλώσει ότι θέλουν να προχωρήσουν ακόμα πιο πέρα όσον αφορά την κλιματική διάσταση στην εξωτερική μας συνεργασία. Σε στενή συνεργασία με συναδέλφους στη Γενική Διεύθυνση για το κλίμα και για το περιβάλλον, για να στηρίξουμε τους στόχους αυτούς, τα τελευταία χρόνια έχουμε αναπτύξει ένα εκτενές σχέδιο κλιματικής διπλωματίας που εφαρμόζουμε σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη. Βρισκόμαστε τώρα πια στην τέταρτη γενιά όσον αφορά το θέμα αυτό. Ε, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε επαφές με εταίρους σε όλο τον κόσμο πριν και μετά από κάθε ετήσια ε, συνάντηση, διάσκεψη των μερών, κάθε COP δηλαδή, ώστε να ενσωματώνουμε τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης σύμφωνα με τη Συμφωνία του Παρισιού στη συνεργασία μας με αυτούς τους εταίρους. Και ακριβώς γι' αυτό τονίζουμε την ανάγκη ενίσχυσης του συστήματος του ΟΗΕ καθώς και την ανάγκη επαρκούς χρηματοδότησης ώστε με τις συνεργασίες μας να μπορέσουμε να πετύχουμε τους φιλόδοξους στόχους που καταγράφονται στη Συμφωνία του Παρισιού. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για την παρέμβασή σας αυτή. Δεν βλέπω να ζητάει κανείς άλλο το λόγο. Θα πρέπει να συνεχιστεί η συνεργασία ανάμεσα στις επιτροπές μας. Θα ακούσουμε κάποια συμπεράσματα από τον πρόεδρο της ΕΝΒΗ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Εγώ δεν είχα πρόβλημα να ολοκληρώνατε εσείς ε, τη συνεδρία. Τέλος πάντων, αυτό που πρέπει πιστεύω να γίνει, να συνεχιστεί αυτή η πρόοδος ε, και ιδίω η διάσκεψη κορυφή τη Νέα Υόρκη θα έχει ζωτική σημασία και από ό,τι γνωρίζουμε θα υπάρξει αντιπροσωπική. Αρχές Σεπτεμβρίου θα κάνουμε την προετοιμασία και καλό θα ήταν ε, να γίνουν τα επόμενα βήματα στη Νέα Υόρκη θα φροντίσουμε να γίνει αυτό. Μας είπε και πριν ε, ε, η μέρη του Μαγκενσκάτ πρέπει να το έχουμε πάντα κατά νου. Οι στόχοι βιώσιμη ανάπτυξη δεν αφορούν μόνο τι αναπτυσσόμενε χώρε, αλλά και εμά του ίδιου. Και νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να το θυμίζουμε συνεχώ στου εαυτού μα. Να μην κοιτάμε μόνο προ τα έξω, αλλά και τα του οίκου μα. Πολλά έχουμε να κάνουμε και εμεί εδώ. Πολλά πρέπει να γίνουν και σε επίπεδο κρατών μελών για την εφαρμογή των στόχων βιώσιμη ανάπτυξη. Και από την προοπτική της ΕΝΒΗ, οι συνάδελφοι της ΝΤΕΒΕ, ξέρω ότι θα συνεδριάσουν και αύριο. Για τους συναδέλφους από την ΕΝΒΗ πρέπει να πω ότι εμείς ε, κλείσαμε και ως ΕΝΒΗ θα ξανασυνεδριάσουμε 4 Σεπτεμβρίου για την προσεχή μας συνεδρίαση. Ωραία. ΝΤΕΒΕ. Εμείς τα λέμε αύριο 9 το πρωί. Ε, έχουμε έτσι μια πλήρη ατζέντα πριν από τις θερινές διακοπές. Μη φοβηθείτε.